<laughs> Domnul președinte. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Το εκτιμώ. Συνεχίζουμε τη σύνοδο. Να ψηφίσουμε τα χθεσινά πρακτικά και τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν είναι διαθέσιμα. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, θεωρώ ότι τα πρακτικά έχουν εγκριθεί. Έχω μια